Άρα στον ετούντον άσυλο. Ο κύριος ε, ο, ο Νίκολας Σμίτ έχει το λόγο. Okay. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, από την αρχή της Προεδρίας μας δεσμευτήκαμε και προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις στην ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε από τις μεταναστευτικές ροές. Ήμασταν αποφασισμένοι να δράσουμε δίχως καθυστέρηση για να βρούμε αποτελεσματικά μέτρα με αλληλεγγύη που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτική που ακολούθησε το Συμβούλιο λοιπόν έχει ως στόχο να συνδυάσει όλες τις προσπάθειες για να προστατεύονται τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία και δικαιούνται εθνικής προστασίας και επίσης στόχος μας ήταν να βελτιώσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να διασφαλίσουμε έτσι την προστασία και την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν μέσα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήματος ασύλου μας. Πρέπει αποτελεσματικά να ανταποκριθούμε στην ανθρωπιστική ανάγκη και να διασφαλίσουμε την διεθνή προστασία, σύμφωνα πάντα με τις υποχρεώσεις μας που έχουμε σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά την κράτηση. Ο βασικός κανόνας του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου είναι ότι κάθε μετανάστης, όπως οποιοδήποτε άλλος, έχει δικαίωμα στην ελευθερία. Η κράτηση δεν μπορεί να είναι παρέκτακτο μέτρο. Δεν δικαιολογείται παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στο κεκτημένο σε σχέση με το άσυλο και τη μετανάστευση και ιδίω στην οδηγία για την επιστροφή και την οδηγία τη σχετική με τις συνθήκες υποδοχής των ετούντων άσυλο. Η οδηγία για την επιστροφή προβλέπει ότι οι χώρες μέλη δεν μπορούν να προσφύγουν στην κράτηση παρά μόνο εφόσον άλλα μέτρα, λιγότερο κατασταλτικά και περιοριστικά, έχουν εφαρμοστεί. Πρόκειται για το άρθρο 15, πρώτη παράγραφος. Κάθε κράτηση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη και δεν μπορεί να παραταθεί παρά μόνο όσο χρειάζεται βάσει της διάταξης η οποία εκτελείται με όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται. Επίσης, η οδηγία σχετική με τις συνθήκες υποδοχής των ετούντων άσυλο προβλέπει στο άρθρο 8 ότι κανείς δεν μπορεί να βρεθεί σε κράτηση απλώς και μόνο επειδή ζητάει διεθνή προστασία. Κράτηση δεν ε, μπορεί να είναι δυνατή παρά μόνο εφόσον είναι αναγκαία και εφόσον κατά περίπτωση εκτιμηθεί και δεν μπορούν να ληφθούν αποτελεσματικά άλλα μέτρα λιγότερο περιοριστικά. Ακριβώς επειδή έχουν διεθνείς δεσμεύσεις οι χώρες μέλη και επειδή υπάρχουν οι κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρε μέλη πρέπει να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αυτών σύμφωνα με τι οδηγίε. Εφόσον δεν εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τις χώρες μέλη, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθηκών πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος επιστροφής, το Συμβούλιο πολλές φορές τους τελευταίους μήνες έχει πει ότι η χρήση της κράτησης δεν μπορεί παρά να είναι το τελευταίο μέτρο και δεν είναι δυνατόν να τίθεται σε εφαρμογή δηλαδή παρά μόνο εφόσον άλλα μέτρα έχουν εφαρμοστεί ή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Στα συμπεράσματα της 9 η Νοεμβρίου το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι χώρες μέλη σε περίπτωση μη συνεργασίας των μεταναστών που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν πράγματι να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το κεκτημένο της Ένωσης. Δηλαδή να υπάρχουν και περιοριστικά μέτρα και ακόμα και κράτηση εφόσον αυτή δεν παρατείνεται περισσότερο από όσο χρειάζεται για να τηρηθούν οι διαδικασίες. Μόνο βέβαια εφόσον τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα από τις αρχές και η αρχή της μη επιστροφής, νόρε φουλμό. Όσον αφορά την μετεκατάσταση 120.000 ατόμων από την Ελλάδα και την Ιταλία, οι χώρε μέλη συμφώνησαν ότι εφόσον σε θελοντική βάση δεν είναι εφικτή μια επιστροφή και άλλα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία για την επιστροφή δεν είναι κατάλληλα, τότε μέτρα κράτησης σύμφωνα με την σχετική οδηγία θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή εκτάκτος. Στα πλαίσια αυτά θέλω να υπογραμμίσω ότι οι μετανάστες δεν έχουν την επιλογή του μέρους προστασίας τους και ότι απαιτείται η πλήρη συνεργασία τους προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα της μετεγκατάστασης. Τέλος, όσον αφορά την χρήση βίας, στα πλαίσια των ε, δακτυλικών ε, από εδώ υπάρχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της 22ης Οκτωβρίου, απόφαση η οποία μιλάει για τους εμπειρογνώμονες επιτόπου. Συνεπώς και αν κατακλείδη. Το θέμα της κράτησης παραμένει ένα σημαντικό θέμα. Μόνο εκτάκτος μπορεί να εφαρμοστεί και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα από κοντά δεδομένου ότι οι διευκρινήσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα αυτό αναμένονται προσεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, Υπουργό και τώρα εκ μέρους της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Μέλη του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται με το Κοινοβούλιο το στόχο της πλήρους συμμόρφωσης των πολιτικών μας με τις ανάγκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ανθρώπινες αξιοπρέπειες. Αυτό βρέθηκε και στον πυρήνα της συζήτησης για την έκθεση που μόλις ολυρώσατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Μιλάμε για μια βασική μέρημνα σε ό,τι αφορά και τους ετούντες άσυλο. Και στρέφομαι τώρα στο θέμα της δήλωσης. Πράτηση και χρήση βίας κατά των ετούντων άσυλο. Το δικαίωμα της ελευθερίας και ασφάλειας ε, των ε, ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων οδηγεί και στο δικαίωμα του ασύλου, που είναι και αυτό θεμελιώδες. Τους περασμένους μήνες, όπως θα θυμάστε, έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να καταφέρουμε σε όλα τα μέτωπα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να γίνεται σεβαστή. Αυτό σημαίνει σεβασμό όλων των πτυχών της νομοθεσίας περί ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο και επειδή υπήρχε και ο έλεγχος μη επαναπροώθησης και αναλογικότητας, οι χώρες μπορούν να ανοιχθούν την είσοδο σε άτομα που δεν έχουν εκφράσει την επιθυμία να ε, υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία. Όπως επίσης γνωρίζετε, έχουμε καταβάλει προσπάθειες για να υπάρχει κατάλληλη καταγραφή των προσφύγων, ασχέτως με το καθεστώς τους. Αυτό είναι προϋπόθεση ώστε να μπορούμε καταλήλως να διαχειριστούμε τις ροές αλλά και τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των μεταναστών. Να αποσαφηνίσω τι απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την οδηγία ΡΙΚΑ στι επαναδιατυπώσει των οδηγιών περί ασύλου που εγκρίθηκαν με συναπόφαση, το κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει σαφεί κανόνε για την κράτηση των ατούντων άσυλων που ε, ορίζουν ένα συγκεκριμένο σημείο ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Είναι λοιπόν ε, καθοριστική σημασία τα πρόσωπα να κρατούνται πάντοτε σε συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες. Εδώ η κράτηση πρέπει να είναι μια έσχατη λύση και μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι εναλλακτικέ της κράτησης. Συμφωνούμε όλοι ότι κανένας δεν πρέπει να, κρατάτε, να κρατείται για τον μόνο λόγο ότι εκείνη ή εκείνος είναι απλώς ετών άσυλο. Όταν ε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ε, διαφυγής θα πρέπει οι μετανάστες να ε, τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης αναλογικά και εφόσον αυτό είναι δικαιολογημένο. Επίσης η οδηγία για, τα, για τις συνθήκες κράτησης προβλέπει ότι οι συνθήκες κράτησης των ετούντων άσυλο Πρέπει να σέβεται όλου του κανόνε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τι ε, βασικέ του ανάγκε. Το να υπάρχει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο είναι μόνο η μισή πορεία που πρέπει να διανύσουμε. Η πραγματική πρόκληση τώρα είναι να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συνεπή και σταθερή υλοποίηση όλων αυτών των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά το πώ τα κράτη-μέλη σέβονται του ευρωπαϊκού κανόνε για την κράτηση. Τα κρατη πρέπει να μεταφέρουν την ε, οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής ως τον Ιούλιο του 2015. Έπρεπε να την έχουν μεταφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιστολή έχει στείλει ειδοποιητήριες επιστολές στα κάτι μέλη που δεν γνωστοποίησαν, δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς που προέβλεψαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης δίνει μεγάλη προσοχή στο τι κάνουν στην πράξη τα κάτι μελη σε αυτό το τομέα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει συμβουλές και καθοδήγηση στα κατημέλη προκειμένου να διευκολύνει την συστηματική λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τους ε, μετανάστες. Και αυτό για να έχουμε καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω της καλύτερης υλοποίησης της οδηγίας Eurodac, ενώ ταυτόχρονα να γίνονται σεβαστά και τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών μέλη του Κοινοβουλίου σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ήθελα να, να ζητήσω την ε, κατανόησή σας κάτι περισσότερο από ό,τι προγραμματιζόταν ε, η προηγούμενη συζήτηση και σε μισή ώρα πρέπει να προλάβω την πτήση για Βερολίνο. Θα με αντικαταστήσει ο Επιτροπός κ. Στυλιανίδης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ και τώρα η εκπροσωπή των πολιτικών ομάδων η κυρία Χολμάγερ από το ΕΛΚ πρώτη. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω για αυτή την σύντομη επισκόπηση. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κράτη-μέλη στα οποία ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων ή των οικονομικών μεταναστών δεν τηρούνται επαρκώς. Ε, δεν έχει σημασία ε, εάν ε, υπάρχει λόγος. Ε, η χρήση βίας δεν επιτρέπεται είτε μέσα στη φυλακή, σε κάποιες δομές που μοιάζουν με φυλακή, γιατί φαίνεται ότι οι συνθήκες εκεί μπορεί να είναι χειρότερες και από φυλακή. Δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη, οι συνθήκε υγιεινή είναι πολύ κακέ. Ε, χρησιμοποιούνται δακρυγόνα. Αυτό μπορεί να είναι στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, σε οποιοδήποτε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που πρέπει εμεί να κρίνουμε είναι ε, ε, η σωστή και με μέτρο αντιμετώπιση ανθρώπων που έχουμε απέναντί μας. μπορούμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε λύσουμε αυτό πρώτα απ' όλα. Η υποχρέωση για την καταγραφή είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική και πρέπει εξ αρχής να το ορίσουμε, ειδικά για τους νέους και τα παιδιά ε, που δεν έχουν ενημερωθεί σωστά από τους ε, λαθρέπορους ε, και δεν έχουν καταγραφεί σωστά ή δεν έχουν καταγραφεί υπό τις σωστές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και ε, λόγω αυτού έχουν γίνει θύματα του εγκλήματος ε, γιατί τα έχουν εκμεταλλευτεί με ε, πολύ άσχημο και βίαιο τρόπο από το αναργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί όλοι και να είμαστε και λογικοί. Ευχαριστούμε την κυρία Χόλο Τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Κεραίρος Σαλόμ. Ευχαριστώ. Αν όλε οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στηρούσαν αυτά τα οποία μας είπαν ο κύριος Σμίτ και ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι η ελευθερία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ότι η στέρηση ελευθερίας είναι κάτι που κατά περίπτωση μόνο μπορεί να γίνει και που πρέπει να αιτιολογείται και ότι μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν μπορούν να επιστρέψουν τότε δεν θα συζητούσαμε σήμερα το βράδυ αυτό το πράγμα. Όμω, δυστυχώ αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν βάλει σειρματόπλεγμα, έχουν φτιάξει τείχη, οι οποίε επιθετικά αντιμετωπίζουν του ετούντε ε, άσυλο, τους πρόσφυγες και υπάρχουν χώρε οι οποίε δεν τηρούν τα δικαιώματα αυτά και ασκούν βία. Μα το θέμα δεν είναι να συμπεριφερόμαστε άσχημα σε αυτούς που ζητούν άσυλο, αλλά να στείλουμε μήνυμα αποτρεπτικό σε αυτούς που ετοιμάζονται να έρθουν, ώστε να μην ζητήσουν άσυλο στις χώρες εκείνες που τους αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό συζητάμε τώρα. Και αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να αλλάξουμε. Το Δουβλίνο δεν λύνει το πρόβλημα. Συμφωνούμε όλοι για το ότι πρέπει να βρεθούν νέες προδιαγραφές που θα μας επιτρέπουν να ρυθμίζουμε αυτή την κατάσταση διαφορετικά. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι οι ανθρωπιστικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν όταν θέλουμε να προστατεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τον πόλεμο όπου κινδυνεύει η ζωή τους ή άλλοι θέλουν να ξεφύγουν από την πείνα που μερικές φορές είναι κάτι πιο βίο ακόμα και από τον πόλεμο. Οι χώρες μέλη λοιπόν πρέπει να φροντίσουν για τη σωστή διαχείριση της πολιτικής μας ασύλου που περιέγραψαν πολύ καλά και το Συμβούλιο και η Επιτροπή αλλά που δυστυχώς πολλές χώρες μέλη δεν τηρούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους των συντηρητικών, ο Τίμωθη για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ήδη το έχω πει πάνω από μια φορά αυτή την εβδομάδα, αλλά η σωστή εφαρμογή των κανόνων που έχουμε ήδη θεσπίσει είναι το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε ενώπιόν μα. Όσο μεγαλώνουν οι προκλήσει, τόσο πιο καλή η εφαρμογή πρέπει να γίνει. Σε ε, πάρα πολλέ περιπτώσει έχω εδώ ε, στο σώμα πει ότι του κανόνε δεν του τηρούμε και πριν έρθει σε εμά αυτή η κρίση. Όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη το κάνουν και ξέρουμε ότι η Κομισιόν θα είχε, έπρεπε να είχε κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι κάνει τώρα για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Κατανοώ ότι η χρηματοδότηση και η δυνατότητα των κρατών μελών να δώσουν τους κατάλληλους πόρους είναι κάτι που αποδεικνύεται πολύ δύσκολο, όμως αυτό δεν πρέπει να μπαίνει στον δρόμο ε, και να μην ε, αφήνει την τήρηση των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την μεταναστευτική κρίση. Ε, η συνοριακή έλεγχη, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η βελτίωση των συνθήκων κράτησης, όλα αυτά είναι ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Ήρθε λοιπόν η στιγμή η Κομισιόν να δείξει στα κράτη-μέλη πως και αυτά πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Θα πρέπει να μπορέσουμε να λύσουμε τα πράγματα που, ε, με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι, κυρίως με τους κανόνες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας πριν πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Έκερ. Θέλετε να την απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλάτε για την ε, μεταναστευτική κρίση η οποία θα μπορούσε να μπει στην άκρη αν είχαμε την ελεύθερη κίνηση ε, που ε, είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση. Ο κύριος Κάμερον είπε στο Bloomberg ότι θα επαναδιαπραγματευτεί αυτό το θέμα και τώρα έχει δηλιάσει. Γιατί παρετήθηκε και έχασε την ευκαιρία να ρυθμίσει αυτό το θέμα μια και καλή. Απάντηση να πω ότι αυτό είναι λίγο αξιολυπητό. Δεν είχα χρόνο να μιλήσω περισσότερο για τα θέματα τα μεταναστευτικά. Είμαι πεπισμένος ότι ο ηγέτης του κόμματός μου και του Ηνωμένου Βασιλείου θα, θα διαπραγματευτεί τα ζητήματα αυτά, όχι μόνο προς όφελος της Βρετανίας, αλλά και των ε, συνόρων μας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λυπηρό ε, που υπάρχει αυτή η παρένοχληση από ακραία κόμματα στη χώρα μου και δεν συμβάλλουν στην πολύ σημαντική συζήτηση που όλοι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Για δύο λεπτά, εκ μέρους των φιλελεύθερων, η κυρία Βίξρο. Η σημερινή συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αρχίσουμε να στοιχειοθετούμε μια συζήτηση που έχει αρχίσει να γίνεται σουρεαλιστική καθημερινά. Το, χαρακτηριστικό, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του κ. Τούσκ, ο οποίος προβάλλει την ιδέα όλοι οι αιτούντες άσυλο να κρατούνται για 18 μήνες προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι ενδεχομένως τρομοκράτες. Και το πιο περίεργο είναι ότι δεν φαίνεται καν να συνειδητοποιεί ότι αυτό θα αντίκει το τελείω με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να το ξαναπώ λοιπόν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει όλες οι διαδικασίες για την αναζήτηση διεθνούς προστασία στην Ευρώπη και την διαφυγή από συνθήκες πολέμου ή διώξης από το μικρότερο βρέφος μέχρι τη γυναίκα πρέπει να οδηγούνται σε τρόπεδα συγκέντρωσης για 1,5 χρόνο. Αυτό κύριε Πρόεδρε σημαίνει ότι περνάμε τις ζωφερότερες στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία που δεν θέλουμε να ξαναγραφτούν ως σελίδες. Είναι ε, είναι πραγματικά ε, αδιαστικό και είναι και αποτρόπαιο. Θα έπρεπε δημοσίως να ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Τούσκ. Επίσης ακούμε να γίνεται λόγος για μετανάστες που παρανόμως παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν είναι μόνο παραπλανητικό, είναι και εσφαλμένο. Δεν μπορούν να μπουν σε μια χώρα οι άνθρωποι αυτοί αλλιώ για να ζητήσουν άσυλο. Είναι αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαιώμα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συνεργαστούμε, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε καταφύγιο σε όσοι το χρειάζονται. Ανταυτού όμως, οι εντυνόμενοι εθνικισμοί έχουν ε, τελικά καταλύσει αυτές τις συζητήσεις από λαϊκιστές και εθνικιστές που δεν θέλουν ευρωπαϊκή λύση αλλά να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να βρεθεί μια λύση είναι να τη βρούμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. you have a blue card colleague. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μια γαλάζια κάρτα όχι εσείς κύριε Μπονάνο. Ο συνάδελφος ε, εκεί, πάνω. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία μου, νομίζω ότι είστε ιδιαίτερα μεροληπτικοί και πραγματικά διασταυρώνετε τα λεγόμενα του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λέγοντας ότι προτείνει τέτοια διαδικασία. Αν δεν σας άρεσε αυτό που πρότεινε, εσείς τι διαδικασία θα προτείνατε δηλαδή να εφαρμόσουμε, διότι κανείς δεν θα δεχόταν αυτομάτως να καλωσορίζουμε όλους τους μετανάστες και να τους χαρακτηρίζουμε αμέσως και ως πρόσφυγες. Εσείς τι προτείνετε για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ευρώπης. Η δική μου πρόταση είναι απλούστατη. Και νομίζω ότι συγκεντρώνει και την πλειοψηφία τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την οποία είμαι συντονίστρια. Κοινή ευθύνη και ανάληψη των ευθυνών. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει με μια κλίδα κατανομή για τα κάτι μέλη, με προσωπικά δεδομένα όπω ο πληθυσμό, το ΑΕΠ, ε, το ποσοστό απασχόληση και ούτω καθεξής. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, το τι γίνεται με τις χώρες που έχουν κάνει τα περισσότερα για τους πρόσφυγες ως τώρα, όπως η Ιδία, η Γερμανία, η Αυστρία και άλλοι. Είναι επιτέλους ώρα οι χώρες που δεν έχουν συμμετάσχει να σηκωθούν και να ανασκουμποθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Διότι σήμερα αυτή είναι η κατάσταση, αλλά αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και όλοι θα είμαστε ισχυρότεροι αν είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου τώρα τη αριστερή ομάδα, 1,5 λεπτό και ο Σχουαρίστια Μπαούντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από ένα μήνα συζητούσαμε με έναν νέο Αφγανό στα σύνορα ανάμεσα στη Σερβία και τη Βουλγαρία. Αφού πέρασε από το Ερά την Τουρκία, ο Μπιλάλ τελικά κατέληξε στην κόλαση τη Βουλγαρία. Και εδώ καταδικάζω τι καταχρήσει που γίνονται σε βάρο των ανθρώπων αυτών προσφύγων και μεταναστών που πέφτουν στα χέρια τη βουλγαρική αστυνομία. Ξύλο, εκβιασμοί, κακοποίηση. Και η Oxfam και η Διεθνής Αμνηστία και η ΑΚΝΟΥΡ καταγγέλουν ακόμα και δαγκώματα από τα σκυλιά της αστυνομίας έχουν διαπιστώσει τους ανθρώπους αυτούς και πληγές και ματώματα. Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα να περάσουν τα δεχτυλικά τους ε, αποτυπώματα στην ε, Βουλγαρία και μετά πήγαν και στην Σερβία από τον Δημητρό αλλά και εκεί τους κακοποίησαν. Τα άτομα αυτά κρατούνται. Τους ξυλοκοπούν, τους κλέβουν χρήματα οι αστυνομικοί και αντικείμενα αξίας. Και μετά βρίσκονται κρατούμενοι με ελάχιστο νερό και τρόφιμα. Έχω εδώ φωτογραφίες των ανθρώπων αυτών σε κάποιο δάσος που ξεκοροζόντουσαν για λίγο και ελάχιστες φωτογραφίες από το κέντρο κράτησης στη Βουλγαρία. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συμβαίνουν με πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά αυτά συμβαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βουλγαρία, βία της αστυνομίας, ε, κακοποίησεις, διαφθορά. Μιλάμε για πάνθρωπες συνθήκες και για μια πολιτική ασύλου που δεν αξίζει αυτό το όνομα. Είναι απαράδεκτα τα γεγονότα αυτά και απαιτούμε να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα γι' αυτά. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Τζαμπάτσκι. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα οι καταγγελίες αυτές δεν είναι αλήθεια. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το Αφγανιστάν δεν είναι Σύριοι, είναι Αφγανοί. Οπότε ρωτάω, πότε είναι η τελευταία φορά που πήγατε στα σύνορα Τουρκίας-Βουλγαρίας να δείτε τι γίνεται εκεί. Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για εξωτερικά σύνορα και δεν βλέπω ότι διαφέρει από το Παρίσι. Οι Αφγανοί θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι είναι άνθρωποι σαν τους Σύριους. Και δεν πρόκειται μόνο για Αφγανούς. Εμείς δεν ε, καταδικάζουμε μόνο αυτή την περίπτωση. Δείτε και την Oxfam και τη Διεθνή Αμνηστία, την Αχνούρ. Δείτε τις δικές τους εκθέσεις που καταγγέλουν αυτή την πραγματικότητα. Δεν είμαστε μόνο εμείς από την ΚΟΕ. Τώρα για δυόμιση λεπτά εκ της ε, ΚΟΕ, ε, κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την άλλη μεριά ε, ακούμε διάφορα για τον Ντόναλτ, ε, τον Ντόναλτ Η αντίδρασή του μετά το Σαν Μπερναντίνο ήταν κάτι που μας εξέπληξε. Έχουμε το δικό μας Ντόναλτ. Υπήρχε ο Ντόναλτ μάλλον στην άλλη μεριά του, του Ατλαντικού, στην Αμερική, για τις αντιδράσεις του μετά από αυτά που έγινε στο Σαν Περναντίνο. Έχουμε και εμείς τον δικό μας λοιπόν Ντόναλτ, τον Ντόναλτ Τάσκ, που κι αυτός είπε κάτι απαράδεκτο, ότι όλοι οι μετανάστες πρέπει 18 μήνες να κρατούνται. Μα εδώ δεν πρόκειται μόνο για τον περιορισμό του, των προσφύγων, είναι και το θέμα της ασφάλειας. Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι δυνατόν για 18 μήνες να κρατείται ένας ε, πρόσφυγας ή μετανάστης. Είναι απαράδεκτα όλα αυτά. Ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλτ Τάσκ αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ότι είναι επικίνδυνοι για την ασφάλειά μας. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει λοιπόν ο άλλος Ντόναλτ και ο δικός μας Ντόναλτ. Ο Τραμπ έχει δημιουργήσει πόλεμο στο ίδιο του το κόμμα. Άνθρωποι από το δικό του το κόμμα διαφωνούν και θεωρούν απαράδεκτα αυτά τα οποία είπε και θεωρούν ότι παραβιάζει το πρώτο άρθρο του Αμερικανικού Συντάγματος. Και ο δικός μας όμως. Ο Κάμερον, ο Ρέντσι, ο Λάντ δεν τα άκουσαν αυτά. Δεν θα έπρεπε να του πούνε, Ντόναλτ, λάθο παράδειγμα δίνει. Δεν πρόκειται για του πρόσφυγε για του μετανάστε. δεν είναι αυτοί οι τρομοκράτε. Πρόεδρε, Εσεί, ξέρετε τον νόμο, εγώ τον ξέρω, ο επίτροπο επίση ο κύριο Σμίτ γνωρίζει ποιο είναι ο νόμος, ο Ντόναλτ δεν το ξέρει. Μα τι λέει ο κύριο Στάς, κύριε Σμίτ, δεν μπορείτε να τον ενημερώσετε. Το Λουξεμβούργο συμφωνεί με αυτή τη δήλωση του Προέδρου του Συμβολίου. Δεν μπορεί να είναι αυτό παράδειγμα να ακούσουμε και μεθαύριο δηλαδή τέτοια αντίστοιχα. Αυτό είναι το δώρο που μας κάνει για τα Χριστούγεννα. Ο πρόεδρος Τούσκ θα πρέπει να αποσύρει αυτά που είπε. Πρόεδρε, ένα είναι σίγουρο. Από τον Τόναλτα στον πρόεδρο του Συμβουλίου δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο χριστουγεννιάτικα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από, τον κύριο την κυρία Άτκισον. Κυρία μου, δεν θεωρείτε ότι ο Ρέντζι, ο Τούσκ, ακόμα και ο κύριος Κάμερουν ακούνε τους ανθρώπους που εκπροσωπούν. Δεν είναι κάτι μαγικό. Ακούν τις ανησυχίες των πολιτών τους και θα σας πρότεινα να κάνετε και εσείς το ίδιο. Πριν απαντήσετε, επειδή δεν είναι ερώτηση, να σας θυμίσω συναδελφοί ότι η μπλε κάρτα είναι για ερωτήσεις και όχι για δηλώσεις. Ε, ίσως ε, η γνώση μου της γραμματικής στα αγγλικά να είναι μικρότερη από τη δική σας, αλλά τέλος πάντων θα απαντήσετε. Το θέμα είναι, η ερώτησή σας μάλλον συμφωνείτε μαζί μου. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Και ο δικός σας ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει αρκετή αξιοπρέπεια να μην λέει ότι πρέπει να κλειδώνουμε όποιον μετανάστη φτάνει στις χώρες μας. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Να μην τρομάζουμε περισσότερο τους ανθρώπους. Εσείς τρόμο παρουσιάζετε εδώ που θα οδηγήσει σε περισσότερη φτώχεια και ακόμα περισσότερο τρόμο. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Και τώρα για δύο λεπτά εκ μέλους του EFTD Diane James. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ένα κομμάτι της λογικής και της συνοχής στην πολιτική μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επανεγκατάστασης έχουν μπει τώρα στο προσκήνιο. Η κυρία Μέρκελ ε, έχει πει τόσα πράγματα και μιλά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, κάποιες από τις, ε, κάποιοι από τους ανθρώπους που έρχονται μπορεί να είναι ειλικρινώς ε, ετούντες άσυλο ή πρόσφυγες, αλλά λένε κάποιοι ότι αυτοί μας καρεύονται και λένε ότι είναι τέτοιοι ενώ δεν είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι τα προβλήματα που η κακή κρίση της κυρίας Μέρκελ δημιούργησε έχουν επιδεινωθεί λόγω αυτού. Έχουν καλυφθεί επίσης ε, στα μέσα ε, περιπτώσεις ε, πυρκαγιών και άλλων τέτοιων περιπτώσεων βίας σε κοινότητες στην Γερμανία και την Σουηδία όπου έχουν εγκατασταθεί μετανάστες. Πραγματικά υπάρχει αυτή η δυσπιστία και δεν ξέρω πόσο κατανοητό είναι αυτό για μια κοινότητα 197 ατόμων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λίγο τι γίνεται. Δεν ξέρουμε μόνο ε, δεν αγνοούμε μόνο τις δικτατορικές πολιτικές αλλά και τον έλεγχο του ασύλου και την, ε, μετεκατάσταση, της επανεγκατάστασης ε, των μεταναστών. Όλα αυτά έχουν συμβεί διότι η πίεση είναι πολύ μεγάλη, περισσότεροι από αυτοί που μπορούν να αντέξουν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μάθει από τα λάθη της και να αλλάξει πλήρως κατεύθυνση. Καλό θα ήταν για να, ομαλοποιήσουμε τη διαδικασία ενσωμάτωσης, να σταματήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις βίας, να σταματήσουμε να φερόμαστε ως δικτάτορες, να πούμε στην κυρία Μέρκελ να κατανοήσει ε, τι ακριβώς λέει και να ε, αλλάξουμε ρότα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, η Βίκη Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χιλιάδες πρόσφυγες βρήκαν το δρόμο τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα τσουνάμι που έφτασε και στη χώρα μου και στην ε, Ολλανδία. Είναι πάρα πολλοί οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει με όλες τις συνέπειες. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Η Ολλανδία είναι ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί. Εγκληματίες ε, δεν πρέπει να έχουν θέση εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όσον αφορά το κόμμα μου, το κόμμα της ελευθερίας, η ασφάλεια των Ολλανδών βρίσκεται πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Οι πρόσφυγες όντως πρέπει να περνάνε από screening για να μην είναι εν δυνάμει εγκληματίες οι τρομοκράτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καθορίζει το κάθε κράτος μέλος και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τους θέλουμε. Πρέπει να έχουμε σύνορα στην Ολλανδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα για δύο λεπτά Μαρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Βουλγαρία αναφέρθηκε παρελειμμένως εδώ. Και η Βουλγαρία έχει βεβαίως μεγάλες ευθύνε ως μία από τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει φροντίσει να έχει διασυνοριακή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και ε, διεθνείς οργανώσεις και πάντοτε βάσει του διεθνούς δικαίου. Εδώ πρέπει να κάνω τέσσερι παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία για τι εκθέσει παρακολούθηση που αποτιμούν τα εθνικά συστήματα υποδοχή. Και η έκθεση που αναφέρουμε ε, και συζητάμε εδώ δεν χρησιμοποιεί αυτή την ενιαία μεθοδολογία. Όσοι ε, εκφωνούν ε, και εξαπολύουν κατηγορίες κατά των αρχών θα πρέπει να αναφερθούν ονομαστικά. Έπειτα, οι βουλγαρικές αρχές ελέγχονται καθημερινά για το κατά πόσον ε, σέβονται τις υποχρεώσεις τους με συγκεκριμένους ε, επιθεωρητές. Τον Φεβρουάριο του 2015 έγινε η απόφαση να γίνουν πέντε επισκέψεις ελέγχου στα σύνορα και δεν βρέθηκε τίποτε το παράτυπο. Και ίσα ίσα η αρχή της μη επαναπροώθησης είναι κάτι που η Frontex το παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που εξετάζουμε τις περιπτώσεις των υπηκών τρίτων χωρών. Πρέπει να δείχνουμε λοιπόν σεβασμό για τους ίδιους τους οργανισμούς μας όπως η Frontex. Έπειτα οι υπηρεσίες των διεκτικών αρχών περνούν από ειδική εκπαίδευση για την ε, ε, διαχείριση των ε, ετούντων ασύλου. Ε, και αυτό σε καθημερινή βάση. Α μην ξεχνάμε τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται. Κατά τρίτον, η επίσημη διαδικασία για την υποβολή αίτηση, ε, ή μάλλον για την προσφυγή κατά ενό κράτου μέλου για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, απαιτεί την ε, συμπληρώση σχετικού εντύπου και την υποβολή του στι αρμόδιε εθνικέ αρχέ. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο να υπάρξει αντικειμενική εξέταση τη κάθε υπόθεση. Και τέλο, εδώ ο ρόλο μα συνάδελφοι είναι καθοριστικό. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, η ΛΥΜΠΕ, αποστέλει επισκέψει ε, για να ε, πραγματοποιήσουν αποστολέ συλλογή στοιχείων σε όλε τι ενδιαφερόμενε χώρε. Όμω, αυτά τα κράτη-μέλη που κάνουν τεράστιε προσπάθειε, καλό θα ήταν να ενθαρρύνονται παρά να επικρίνονται διαρκώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Βάιντενχολτ για δύο λεπτά. Το μικρόφωνο. Το 2015 ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ένα έτος στο οποίο είχαμε τη μεγαλύτερη κίνηση προσφυγών από ποτέ και δεν έχει περάσει αυτό. Ε, έχουμε ζήσει πάρα πολλά τρομακτικά πράγματα, έχουμε ζήσει ε, ζητήματα ε, με προβλήματα στη Μεσόγειο κτλ. Εδώ και καιρό Μιλάμε όμως για μια ολιστική προσέγγιση και να υπάρχει και μια διαφοροποίηση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την κάθε κατάσταση γιατί ε, υπάρχει, είναι άλλο η μετανάστευση, άλλο το άσυλο, άλλο ο εκτοπισμός. Χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία. Και το πρόβλημα της διαδικασίας ασύλου είναι ακριβώς ότι πρέπει να δώσουμε προστασία, να έχουμε συγκεκριμένη ατομική εξέταση και να εγγυόμαστε σωστές διαδικασίες. Ε, πρέπει να κοιτάμε πάντοτε ε, ποιες είναι οι συνθήκες όταν έχουμε θύματα, έχουμε οδηγίες, έχουμε στάνταρτ που μας καθοδηγούν ε, για να μπορούμε να προστατεύουμε νέους και παιδιά όπως είπαμε. Και, και αναρωτιέμαι ακριβώς γιατί αυτό το πακέτο δεν έχει εφαρμοστεί στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν αυτές τις διαδικασίες, ε, ε, ενώ είναι λογικό και πρακτικό να γίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος, οι legal avenues όπως λέγονται, και να υπάρχουν και τα εργαλεία και ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και με την Τουρκία που αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα. Γιατί ε, ως τώρα δεν το κάνουμε, είναι προβλήματα αυτά που έχουμε στη σχέση μας με την Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα η Χέλγκα Στίβενς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά την επίθεση στο Παρίσι, ο Πρόεδρος τους είπε ότι οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να κρατούνται όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να ελεγχθεί η ταυτότητά τους. Δυστυχώ, κάποιοι από τους υπεύθυνου για τι επιθέσει στο Παρίσι μπήκανε με ψεύτικη ταυτότητα οι μετανάστες δεν είναι τρομοκράτες, αλλά κάποιοι τρομοκράτες μπαίνουν από τα Βαλκάνια, όπως μπαίνουν και πάρα πολλοί μετανάστες. 30% των ε, μεταναστών έρχονται από την Συρία. Πραγματικά μας ε, σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν ε, παράνομα οι μετανάστες και μας σοκάρει αυτό που είπε ο κ. ότι θα κρατούνται. Όμως, πώς θα ελεγχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καλύτερα είναι να ρωτήσουμε γιατί τα εξωτερικά μας σύνορα είναι σαν σουρωτήρι και γιατί η Ελλάδα και η Ιταλία δεν καταφέρουν να εφαρμόσουν τους κανόνες και γιατί η Επιτροπή στρίβει το βλέμμα αλλού και δεν κοιτάει αυτά τα προβλήματα. Αυτά είναι που κάνουν την πληγή να παραμένει ανοιχτή. Η κυρία Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ. Πώς είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να πρέπει ακόμη να εξηγούμε στα κράτη-μέλη, στο λίκνο της δημοκρατίας του κόσμου, ότι δεν είναι νόμιμο τα παιδιά να μπαίνουν στη φυλακή. Παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από φρικαλαιότητες που κανείς από εμάς που δεν γνωρίζει ποτέ. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο το δικαίωμα της ελευθερίας, της προστασίας κατά της ε, αυθαίρετης ε, κράτησης είναι θεμελιώδη δικαιώματα και αναφέροντας την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ισχύουν για κάθε ανθρώπινο πλάσμα χωρίς καμία καμία εξαίρεση. Και όμως διαπιστώνουμε όλο και συχνότερα και μόλις τώρα ακούστηκε ότι οι πρόσφυγες πολλές φορές ε, κρατούνται και κάποιες εκθέσει μιλούν για βασανιστήρια, για μετιστικέ κρατήσεις, για βίες πράξεις. Εδώ λοιπόν συνάδελφοι εξηγήστε μου πώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Τούσκ που ε, μας εκπροσωπεί όλους μπορεί πριν από λίγες μέρες ε, μόλις να δηλώνει ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να κρατώνται, να ως, 18 μήνες τη στιγμή της άφεξής τους στην Ευρώπη. Προκειμένου λοιπόν να μην ταπεινώσουμε και να μην υπονομεύσουμε τελείως τις αξίες μας και να αποδείξουμε ότι σεβόμαστε τα θεμέλια δικαιώματα που τόσο πολύ ε, ζητοκραυγάζουμε σε όλο τον κόσμο ότι προστατεύουμε, καλό θα ήταν να έχουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορα. Να έχουμε κατά κατανομή των ευθυνών. Αυτό είναι ανάγκη. Η αξιοπρέπεια πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλου, στην κάθε μια και τον καθένα, και στον ευρωπαϊκό χώρο και πέραν αυτού. Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλου. Επόμενη κυρία Πιόρκ για μισή λεπτά. Για ενάμιση λεπτό, συγγνώμη. Ευχαριστώ, μαζί με την ε, ε, αντιπροσωπεία της ομάδας της Συνοτικής Αριστεράς πήγαμε στα Βαλκάνια και συναντήσαμε σε διάφορους σταθμούς των σύνορων και αστυνομικούς και συνεροφύλακες και ανθρώπους που προσπαθούσαν ε, να περάσουν τα σύνορα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε κανείς από μας να γνωρίσει. Πραγματικά τους αξίζει μια καλύτερη υποδοχή στην Ευρώπη δεν είναι παράνομοι και δεν θα έπρεπε να τους κλειδώνουμε, να τους ε, φυλακίζουμε και να πέφτουν θύματα βίας. Όμως βλέπουμε ότι στην Τουρκία ήδη τους έχουν συμβεί πολλά δυσάρεστα. Έχουμε σχετικά ε, ε, δε, νέα και ειδήσει. Οι νέοι έχουν περάσει από τέτοιε συνθήκες υποδοχής που θεωρούν ότι έχουν φυλακιστεί. Έχουμε ακούσει βίες, βιαιότητες από την αστυνομία ε, για διώτες από την αστυνομία στην Βουλγαρία. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου είναι τι θα κάνετε για να το πάψετε αυτό το φαινόμενο. Τι θα γίνεται με τις αστυνομικές δυνάμεις των κρατών μελών ε, που κλέβουν τα ελάχιστα υπάρχοντα των προσφύγων και χρησιμοποιούν βία γι' αυτό. Θα στρέφεται την πλάτη αδιάφορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κατημέλη μελη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κανόνες του Δουβλίνου. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα τέτοιας βίας. Θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση, διότι αν δεν κάνετε τίποτα, αντί να μιλάμε για την διεθνή προστασία, ουσιαστικά θα συνεχίσουμε την παροχή βίας και αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να είναι τραυματισμένοι από τις εμπειρίες τους. Κυρία μου, κυρία Μπιόρκ, υπάρχει μια ερώτηση για σας. Τη δέχεστε. Υπάρχει μια ερώτηση για σας. Από τον κύριο Μπονάνο. Όχι, γιατί απλώς θα χαθεί ο χρόνος μου και των συναδέλφων. Η κυρία Κέλλερ, για ένα λεπτό. είναι δικαίωμα των βουλευτών βάσει του ιστορικού να αποδεχτούν ή όχι την ερώτηση. Αν κανείς δεν θέλει, είναι ελεύθερος να μην τη δεχτεί. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ε, κοίταξα το βιογραφικό, ε, μάλλον ε, την περιγραφή της θέσης του κυρίου Τούσκ που υπάρχει στο διαδίκτυο και λέει ότι πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή και τη συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν κοιτάζει αυτή την περιγραφή της θέσης εργασίας του πολύ συχνά και την ιστοσελίδα του. Έπρεπε μάλλον να το κάνει γιατί αυτό που έδωσε στις εφημερίδες δεν βοηθούσε από αυτή την άποψη. Ο πρόεδρος τους και επίσης δεν φαίνεται να είναι πολύ στεναρός όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί ζητά κάτι που παραβιάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Βέβαια, δεν είναι αυτός ο θεματοφύλακας των συνθήκων, αλλά η Κομισιόν. Ο κύριο Γιούγκερ λοιπόν πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του με τον κύριο Τούσκ και στο μέλλον έχουμε πιο συνενετική προσέγγιση και τα θέματα που παρουσιάζει ο πρόεδρο του Συμβουλίου να γίνονται με ένα πιο... Ε, Ευχαριστούμε κυρία Φεράρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόκληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι να καταφέρει να βρει τη σωστή ισορροπία και να εξισορροπήσει ελευθερία και ασφάλεια. Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι εργαλείο. Εργαλείο για να φτάσουμε στην ελευθερία και να βεβαιωθούμε ότι η ελευθερία προστατεύεται ω θεμελιώδη δικαίωμα. Σήμερα όμω φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια εξισορρόπηση ε, ουσιαστικά ε, οδηγεί βάρο τη ελευθερία στην πράσπιση μόνο τη ασφάλεια. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των, των άσυλο, αλλά εις βάρος ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών που τους υποδέχονται και των ε, άλλων πολιτών τρίτων χωρών που νομίμως ζητούν να τους δεχτούμε. Ποια είναι η λύση λοιπόν. Λύση δεν είναι η χρήση βίας βεβαίως, ούτε η διοικητική οδός. είδαμε στην Ιταλία που είναι ένα από τα χειρότερα παραδείγματα των κέντρων επιστροφής και των κέντρων κράτησης να υπάρχουν συνθήκες δυστυχώς πολύ αρνητικές για τη διαβίωση των ε, προσφύγων που φτάνουν ως εκεί. Το κίνημα Cinque Stelle, πέντε αστέρες, θέλει να αναθεωρηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις, οι ανθρωπιστικοί διάδρομη και οδοί. Όλα αυτά είναι λύσεις που έχουν ακουστεί και προηγουμένως και θα πρέπει να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια και για τους ευρωπαϊκούς πολίτες και για αυτούς που δεχόμαστε στην επικρατεία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Μπιτζότο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για μετανάστευση στην Ευρώπη, λέμε πάντοτε τα ίδια. Υποδοχή, αλληλεγγύη, ένταξη. Και ε, συνοπτικά η Ιταλική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να δεχτεί όλους τους λαθρομετανάστες που μόνο μικρό μέρος είναι πρόσφυγες. Και τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα επενούμε την Ιταλία που υποδέχτηκε τόσε εκατό εκατομμύρια πρόσφυγε και μετά τι επιβάλλουμε πρόστιμα διότι δεν μπορεί να ε, διαχειριστεί όλη αυτή τη μεταναστευτική ροή. Ντροπή σα, ντροπή σε όλου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ιταλική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα κέντρα αυτά δεν τα ορίζει, δεν τα ιδρύει στην Αφρική για να ξεκινάμε από την αρχή να διαπιστώνουμε αν υπάρχει καθεστώ πρόσφυγα στον καθένα που ζητάει άσυλο. Και γιατί να φτάνουν όλοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κινδυνεύουν στη θάλασσα θύματα των εμπόρων ε, ανθρώπων φτάνοντα στην Ιταλία. Και γιατί ανήκαν η Ιταλική κυβέρνηση να πρέπει να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κύριε Επίτροπε, η στρατιώτα της Ιταλίας δεν θα ε, χρησιμεύσει τίποτα. Ε, ίσως ε, τους που είναι πιθανοί τρομοκράτες θα τους ε, εντοπίσει. Όμως όχι αυτούς που προσπαθούν να, ξεφύγουν από τον πόλεμο. Σκεφτείτε πόσοι Ιταλοί χρειάζεται να ε, επιζήσουν με ελάχιστα εκατοντάδες ευρώ το μήνα ενώ όλα τα έχουν δωρεάν οι πρόσφυγες. Με κινητά, με στέγη, ε, λες και έχουν έρθει διακοπές. Όχι και πάλι όχι. Ευχαριστούμε κύριο Ζάντεφ για Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σε πολλές εκθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει ότι η Βουλγαρία προστατεύει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα με την Τουρκία αντιμετωπίζουν βέβαια δυσκολίες και είναι δύσκολο να διαπραγματευτούμε. Η αστυνομία στη Βουλγαρία εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ε, βέβαια διαλύει εγκληματικά δίκτυα, συλλαμβάνει ενδυνάμει εγκληματίες και παράνομους μετανάστες και άλλους που πρέπει να τους προστατεύσει, τους προστατεύει. Κακώς κατηγορείται από ξένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις η Βουλγαρία για καταχρήσεις σε βάρος των ετούντων άσυλο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι καμία από τις έρευνες που έχουν γίνει δεν στηρίζουν τις κατηγορίες αυτές. Η παράνομη διέλευση των συνόρων έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούν να μπαίνουν στις χώρες μας, στη Βουλγαρία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εγκληματίες. Γι' αυτό και η Βουλγαρία παίρνει και θα συνεχίσει να παίρνει τα μέτρα που χρειάζονται και που επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να ελέγχει την ροή των παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Θέλω να κάνω έκκληση σε όλους όσοι κατηγορούν τη χώρα και τις χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπείτε στη θέση των συνοριοφυλάκων αυτών πρώτα, πριν μας κατηγορήσετε. Μιλήστε με τους ανθρώπους εκείνους που καθημερινά συναντιούνται με χιλιάδες ε, του Ντεσάσιλο και μετά γράψτε τις εκθέσεις σας. Ε, Ιώτοβα, Δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το 2013 συλλέξαμε διάφορα έγγραφα. Δεν ε, σταματάμε να συζητάμε για την κρίση, αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της κρίσης. Πάρα πολλές συγκρούσεις, πόλεμοι, μας κάνουν να ξεχνάμε τις ανθρώπινες ιστορίες, την ανθρώπινη τραγωδία. Τίποτα όλα αυτά όμως δεν θα είχε συμβεί αν τα μέτρα που προτείναμε ήδη αρχές της χρονιάς είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Οι χώρες μέλη έχουν αποτύχει, έχουν μείνει στην τύχη τους. Και τι κάνουν, βάζουν σειρματόπλημα. Το Δουβλίνο, μα δεν λειτουργεί πια. Οι μηχανισμοί που ίσχυαν δεν ισχύουν πια. Τα hot spots δεν ε, αποφέρουν τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Και δεν είναι σαφή και τα κριτήρια με τα οποία φτιάχτηκαν. Σήμερα ακούσαμε και τη νέα ιδέα 80.000 Σύριοι να μετεκαθίστανται κάθε χρόνο. Ναι, αλλά οι πρόσφυγες δεν είναι δυνατόν να ζουν στην περιφέρεια της Ευρώπης. Φυσικά και προσπαθούν να περάσουν στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Όλα αυτά δημιουργούν εντάσεις. Και θέλω να πω κάτι σε αυτούς που αναφέρθηκαν στη Βουλγαρία ξανά και ξανά. Το μήνυμα σας σήμερα δεν θα πρέπει να είναι να καταδεικνύετε τη μία την άλλη χώρα. Αντίθετα, θα έπρεπε ενωμένοι να αντιμετωπίζουμε τι δυσκολίε. Δεν πρόκειται για κατάχρηση, για βία όταν πρέπει κανεί να πάρει τα δεκτυλικά αποτυπώματα κάποιου ή να βρει την ταυτότητά του. Αυτέ είναι προδιαγραφέ για τι οποίε όλοι ψηφίσαμε. Και όταν μια χώρα όπω η Βουλγαρία ακολουθεί αυτού του κανόνε, δεν πρέπει να την κατηγορείται ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και υπάρχουν μελέτε κάθε χρόνο για το πώς αντιμετωπίζουν την προσφυγική κρίση οι χώρες και δεν έχει κατηγορήσει καμία τέτοια έκθεση τη Βουλγαρία για παραβιάσεις. Όταν λοιπόν μιλάμε με ονόματα, κατονομάζουμε συγκεκριμένες χώρες, αυτό βοηθάει μόνο όσους είναι κατά της Ευρώπης. Σαμπάσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε άλλη μια άχρηστη συζήτηση με μια σωρία εκθέσεων, με λασπολογίες και ψεύδι. Πραγματικά, κατηγορηματικά τα απορρίπτω όλα αυτά μόνον άνθρωποι κακόπιστοι ή που δεν έχουν δει ποτέ τα σύνορα μπορεί να γράφουν τέτοια πράγματα ή δεν έχουν ιδέα για τα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Δεν είναι μόνο τα σύνορα της Βουλγαρίας έτσι, είναι εξωτερικά σύνορα της Ένωσης αυτά. Η Βουλγαρία έχει καθήκον να τα προστατεύει τα σύνορα αυτά για το συμφέρον ε, και την ασφάλεια των βούλγαρων πολιτών και όλης της Ευρώπης, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που μου προσελκύει την προσοχή σε αυτή τη συζήτηση. Ένας, λένε και μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων δεν καταλαβαίνουν τι συζητάμε εδώ πέρα. Μας λένε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όποιος θα μπορούσε να λάβει, μάλλον η λήψη τακτηλικών αποτυπωμάτων είναι, είναι μορφή βίας. Τι πράγματα είναι αυτά. φαίνεται κάποιοι να μιλάνε για αυτού που υποφέρουν, λες και έχουν ε, το σύνδρομο της διχασμένης προσωπικότητα. Τι θέλετε να προστατεύουμε τους λαθρομετανάστες, να τους πάρετε στα σπίτια σας. Ευχαριστούμε γαλάζια κάρτα για σας. Τη δέχεστε. Ο Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σα ρωτήσω, συμφωνείτε ότι οι καταγγελίες γίνονται κατόπιν παρότρισης κάποιων κοιό... και δικηγόρων που κερδίζουν εις βάρος των μεταναστών και που θα έπρεπε να ελεγχθεί ο ύποπτος ρόλος τους. Απαντήστε κύριε Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως θα δείτε, δεν φοβόμαστε να απαντούμε σε ερωτήσεις. Ναι, το πιστεύουμε. Υπάρχουν οργανώσεις που εξυπηρετούν απότερα κίνητρα και συμφέροντα. Και μάλιστα θα ήθελαν η καγκελάριος Μέρκελ να είναι με το πέρας τους. Ευχαριστούμε κυρία Μλίνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Με ανησυχεί το γεγονός ότι ενοχοποιούμε ε, τους μετανάστες. Όταν δεν υπάρχουν νόμιμες δυνατότητες, το να περάσει κανείς παράτυπα τα σύνορα δεν είναι λάθος, δεν είναι έγκλημα, δεν είναι ποινικό αδίκημα και δεν πρέπει κανείς να διώκεται. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο όταν κανείς ζητά το άσυλο και πρέπει να γίνει για να μπορέσει να ταυτοποιηθεί και να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Έχουμε ε, γενικώ ε, ε, να κάνουμε με ανθρώπους και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και παιδιά. Ο τρόπος αντιμετώπισης βέβαια προκαλεί κάποιο κόστος και πρέπει γι' αυτό να, προσέχουμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται σε εμά να μην έχουν ένα ποινικό υπόβαθρο. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την ε, σωστή ε, αντιμετώπιση των προσφύγων. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει μιλήσει για τα hot spot της Ιταλίας και ότι η Ρώμη θα πρέπει να βρει νομικό πλαίσιο για τη χρήση βίας με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αποφυγή μακροχρόνιων ε, φυλακίσεων ή κρατήσεων. Είναι δύσκολο να μην δούμε ότι δύο άρθρα του συντάγματος παραβιάζονται ήδη με αυτές τις προτάσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε κρατήσεις και διεπράξεις κατά των προσφύγων που ε, ολοένα και περισσότερο εξαπλώνονται. Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πολωνία, Γαλλία, Ισπανία, στην Ιταλία, οι βίαιες προσαγωγές γίνονται ακόμη και όταν οι δικαστές δεν δέχονται τον επαναπετρασμό. Οι Δανείοι, οι Βενέζικες αρχές κατάσχουν τα κοσμήματα των προσφύγων με τα οποία τους αναγκάζουν να πληρώσουν το κόστος ε, της μετακινησής τους. Πρέπει να λάβετε μέτρα κατεπηγόντως και να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ. Ο πρόεδρος Τούσκ μιλά για 18 μήνες κράτησης των προσφύγων και για να σώσουμε το Σέγγεν με κάθε κόστος. Δεν είναι όμως υποχρεωτικές οι μη επανοπροωθήσεις. Το χάμπεας κόρπους, οι μη ίδιες ενέργειες κατά ανηλίκων και παιδιών. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μόνο καταστηλτικά μέτρα εδώ, ενώ η χάρτα ε, για τα δικαιώματα των θεμελιών τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι δεσμευτικές μας ε, υποχρεώσεις. Όχι όλα αυτά λοιπόν στο βωμό του Σέγγεν. Ως πολίτης μπορώ να αποποιηθώ το Σέγγεν χωρίς κανένα δισταγμό. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη, η κυρία Ζολή για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Φαίνεται το δράμα των προσφύγων να μην συγκινεί κανέναν και μάλιστα ο πρόεδρος του Συμβουλίου με τις δηλώσεις του υπέρ της ασφάλειας είναι επικίνδυνος και φαίνεται να είναι ένας από τους πολλούς με τη λαϊκιστική φωνή που ακούμε παντού στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι μας σοκάρει περισσότερο. Ότι ο κύριος Τούσκ μπορεί να μιλά για τη δυνατότητα κράτησης των προσφύγων για 18 μήνες για λόγους ασφάλειας ή ότι η πρασινη που ζητούν εξηγήσει για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο δεν έχουν το δικαίωμα να υποβαλούν την προφορική αυτή ερώτηση γιατί δεν συμφωνούν οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε. Το να Αυτά λοιπόν δεν έχουν κανένα νόημα όσο και να τα συζητάμε. Για του πρόσφυγε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να προτείνουμε, ό,τι και να προτείνουμε, βλέπουμε να ε, πέφτουν οι τύχοι αλλά διαρκώς να σκάβουμε νέες τάφρους. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα που στέλνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τέλο το διεθνέ δίκαιο, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη. Μιλάμε μόνο για σύνορα, ασφάλεια και πόλεμο πλέον. Και ποινικοποιούμε ακόμη και περισσότερο τους μετα... όλο και περισσότερο του μετανάστε. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζεται από το διεθνέ δίκαιο. Ιδού η Ευρώπη του 2015. Σα το λέω σήμερα και πραγματικά θα πρέπει να ξεπεράσουμε τι ευχέ και του ευσεβεί πόθου. Θα πρέπει η Ευρώπη να ξαναβρει τη σωστή πορεία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς η κράτηση και η βία είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη δεν έχουν λόγους ε, ε, για να το κάνουν αυτό εύλογους. Και πολλοί άνθρωποι κλέβουν, ε, δηλαδή κάνουν απάτη για να μπουν στην Ένωση δεν θέλουν να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και τα λοιπά, κάνουν ε, σαμποτάζ στη διαδικασία μας. Και στην πραγματικότητα δεν ζητούν το άσυλο από εκεί που θα έπρεπε. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κρατούμε αυτούς τους ανθρώπους και να χρησιμοποιούμε και τη βία, τη βία να ε, χρησιμοποιούμε την ε, μία εθελούσια επιστροφή τους και να χρησιμοποιούμε και το απαραίτητο επίπεδο ε, δύναμης ισχύω ώστε να μπορέσουμε να τους θέσουμε υπό έλεγχο. Νομίζω ότι αυτοί που εκμεταλλεύονται τα συστήματά μας πρέπει να πιάνονται και η χρήση της ε, ε, ισχύω πρέπει να είναι κομμάτι της εργαλειοθήκης που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτούς που κλέβουν. Η κυρία Άτκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δω περισσότερε κρατήσει ειδικά στο Καλέ, γιατί βλέπουμε συνεχώ επιθετικού μετανάστε, κάποιοι με υπόβαθρο τζιχαντιστή, να ε, επιτίθενται σε καθημερινή βάση στου αστυνομικού προσπάθων να κάνουν ε, τη δουλειά του. Ακούμε ε, πολύ μεγάλε φρικαστικέ ιστορίε για φορτηγατζίδε που απειλούνται με μαχαίρια. Εκατοντάδε μετανάστε που φτάνουν στην Νορβηγία έχουν βρεθεί με φωτογραφίε φωτογραφίες ε, τζιχαντιστών στις ε, φωτογραφικές τους μηχανές. Ποιος τους ελέγχει στην ζούγκλα του Καλέ. Πού είναι οι αρχές ε, που θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών μας. Πρέπει να ε, ρισκάρουν τη ζωή τους πριν οι αρχές λάβουν την κατάλληλη δράση. Ε, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπει ο στρατός ε, για να διασφαλίσει την ασφάλεια όπως γίνεται στην υπόλοιπη Γαλλία. Αν μπορούσαμε να βρούμε μια καλύτερη λύση για τη ζούγκλα του Καλέ θα την είχαμε βρει. Γι' αυτό πρέπει να συλλαμβάνουμε, να κρατούμε και να απελάβουμε αυτούς τους ανθρώπους πριν είναι αργά. Για ένα λεπτό, κύριο Σικόφσκα. Δύο λεπτά διορθώνει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους που συζητάμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Δείχνει και αντικατοπτρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις κοινωνίες μας. Δεν συμφωνούμε μεταξύ μας. Δεν βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει μία και μόνη αλήθεια. Είναι σημαντικό όμω το τι άποψη έχει ο καθένας μας. Πριν όμως αρχίσουμε να τα βάζουμε με τον έναν με τον άλλον, καλό θα ήταν να παραδεχτούμε ότι όλοι μας έχουμε σφάλει. Ότι όλοι έχουμε παραβιάσει τους κανόνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μόνο όταν το παραδεχτούμε αυτό όλοι, από εκεί και πέρα μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις στο προσφυγικό. Μιλάμε για την φρικτή κατάσταση των ε, ετούντων άσυλο που περιμένουν στα εξωτερικά μας σύνορα ή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάστασή τους όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί όμως. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι κάνουν. Αυτοί τηρούν όλους τους κανόνες. Θα μπορούσα να μιλήσω για ώρες από την εμπειρία που έχω από προσφυγικούς καταβλισμούς στα σύνορα. Έχουμε ακούσει πολλά για αυτά. Πολλά έχουν υποθεί. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να παραβιάσουν τους κανόνες, να τους παραβούν, που δεν θα προσαρμοστούν και συμμορφωθούν στις διαδικασίες. Είναι ένα θέμα λοιπόν που συζητάμε και καλώς, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλες τις απόψεις. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητάω να μην είσαστε μόνο επικριτικοί. Ας καθίσουμε όλοι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θετικά αυτή την κατάσταση προς όφελος των ανθρώπων εκείνων που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Ο κύριος Ωάννη για δύο λεπτά. Παρακαλώ, Μπορώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στο σώμα και μάλιστα όχι μόνο εδώ. Γενικά στο κοινοβούλιο εδώ γύρω είναι καλό που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Η συζήτηση βέβαια είναι περίπλοκη και δύσκολη. Αν διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης, διαβάζουμε βέβαια αποκλίνουσες απόψεις, διαφορετικές. Όμως, ερευνούν οι... ερευνούμε καταστάσεις που προκαλούν διάφορες κυβερνήσεις όπως η Ουγγρική, που μας ξενίζουν. Υπάρχουν δηλαδή κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν κοινοτικά κονδύλια με τα οποία κάνουν κυβερνητική προπαγάνδα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση των χωρών τους και κάνουν τον κόσμο να τρομάζει. Του λένε ότι βρίσκονται υπό απειλή. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να τηρούμε όλοι τους κανόνες, να φροντίσουμε να εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες και να αποφεύγεται η προπαγάνδα θέλω να αναφέρω κάτι και για το PNR, τους ε, καταλόγους επιβατών. Δεν είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι πολίτες να περνάνε από ένα σωρό ελέγχους για την ασφάλεια και να τηρούν κανόνες και ξανά κανόνες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να διασχίσουν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Εγώ έχω δει ανθρώπους να μπαίνουν και να βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Συνεπώς πρέπει να υπάρχουν ομοιόμορφοι κανόνες που να τηρούνται από όλους. Ευχαριστώ. Χάλα αχώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα από τα βασικά προβλήματα της μεταναστευτικής μας πολιτικής είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να επιστρέψει τους ανθρώπους που οι αιτήσει ασύλου, του έχουν απορριφθεί, έχουν, ασύλου τους έχουν απορριφθεί στις χώρες τους. Αυτό ενθαρρύνει την χρήση του συστήματος ασύλου ως ένα τρόπο οικονομικής μετανάστευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ετούντε περιμένουν σε ανοιχτές και ελεύθερες εγκαταστάσεις την εξέταση της αιτήσή ε, τους και όταν μάθουν ότι απορρίφθηκε εντωμεταξύ συχνά έχουν εξαφανιστεί και παραμένουν, ε, διαμένουν παρανόμως στο χώρο του Σέγγεν ως λαθρομετανάστε. Πολλές φορές εξαφανίζονται τα κέντρα υποδοχής πριν καν καταγραφούν και ληφθούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Όλα αυτά υπονομεύουν την αξιοπιστία του συστήματο ασύλου και θα ήταν καλή ιδέα όλοι μας τους ετούντες άσυλο να φροντίσουμε να τους ε, παρακολουθούμε όσο η υπόθεσή τους εξετάζεται. Αν αυτή δεν είναι ισχύουσα νομοθεσία να την αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστούμε η κυρία Παγκαζαρτουντούα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι γονείς του Ιησού έφυγαν από την Αίγυπτο διωκόμενοι κυρία Βιντζότο, Άτκισον ε, λοιπά πρέπει να το ξέρουν ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάστηκε να φύγουν και γέννησε η Μαρία και αν δεν είχε προστατευτεί ως μετανάστρια θα είχε πεθάνει το παιδί της. Επιτροπή και Συμβούλιο λοιπόν. Δεν υποψιάζεστε καν τι σημαίνει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εσείς θα φταίτε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τον πόλεμο Σήμερα ο κύριος Γιούνκερ τι μας είπε. Μας είπε ότι εμείς γράφουμε την ιστορία. Και αυτή την ιστορία πρέπει να προσέξουμε. Εγώ δεν θέλω να είμαι συνένοχος στην ιστορία που γράφετε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άντερσον. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να πούμε κάτι το οποίο να γράφεται στη βάση του αγάλματος ελευθερίας. Ότι βρίσκομαι εδώ πέρα προκειμένου να αποδεκτώ όλα αυτά τα πλήθη. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα πρέπει και εμείς να εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι οι εθνικές αρχές καλούνται πολλές φορές να κρατούν τους ετούντες άσυλο προκειμένου να προστατεύσουν το αποτυχημένο σύμφωνο του Δουβλίνου και βλέπουμε ότι κινητοποιούν κάποιες ε, ομάδες έκτακτης ανάγκης της ε, Frontex. Πολλές φορές καταπατώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χθε η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της ε, στρέφεται κατά της Τουρκίας η οποία παράνομα κρατά και έχει κακομεταχειριστεί πάρα πολλού ετούντε άσυλο. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει πολλέ φορέ και στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε μία εισβολή. Οι ετούντε άσυλο είναι άνθρωποι σαν και εσά, σαν και εμένα, που μαζί με τα παιδιά του προσπαθούν να διαφύγουν απεγνωσμένα από ένοπλε συγκρούσει στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Πολλές φορές φεύγουν, διαφεύγουν από τους ίδιους συμβαρδισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Από το 1892 το Ellis Island στις Ηνωμένε Πολιτείες έχει προσφέρει ασφαλή είσοδο σε πάρα πολλούς ε, ετούντες άσυλο, σε πάρα πολλούς μετανάστες. Ο Edwin Brock, ένας Ιρλανδός φιλόσοφος, είχε πει ότι το μόνο που χρειάζεται, χρειάζεται για, τη θρία, για τον θρίαβο του κακού είναι οι καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα. Μόνο τότε θριαμβεύει το κακό. Ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακαλώ πολύ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Σας έδωσα κάποια παραπάνω δευτερόλεπτα, αλλά πιέζει πολύ ο χρόνος. Χαουτάλα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία των κρατών μελών προκειμένου να καταφέρουμε να βρούμε ανθρωπιστικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι μετανάστες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε και περισσότερες συμβουλές στα κράτη-μέλη στην εθνική τους πολιτική. Η κράτηση ετούντων άσυλο για περίοδο 18 μηνών όχι μόνο αντιβαίνει στην κοινοτική νομοθεσία, αλλά αντιβαίνει και στο διεθνές δίκαιο. Το να κρατούμε τους ε, τούντες άσυλο σε ειδικά κέντρα ουσιαστικά είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό για τους ίδιους αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να αντιδρούμε με τρόπο λαϊκίστικο, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ενιαία προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης. Ευχαριστούμε πολύ. Σας έδωσα κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω. Ο κύριος ε, Μπέι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Δέκα χρόνια μετά τις τρομοκρατικές, δέκα μέρες με συγχωρείτε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 13 Νοεμβρίου, δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευκόλυναν την καταβολή προσφυγών από τους ετούντες άσυλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι θα έχουμε 3 εκατομμύρια νέους ελαφρομετανάστες μέχρι το 2017 και βλέπουμε ότι δεξιά και αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν στις 2 Δεκεμβρίου ένα ψήφισμα το οποίο ενθαρρύνει τελικά την παράνομη μετανάστευση. Το κείμενο αυτό έχει ως στόχο να εμποδίσει τις συνοροφυλακές από το να κάνουν τη δουλειά τους, δίνοντας κίνητρα κίνητρα στου ε, λαθρομετανάστε για να υποβάλουν προσφυγέ. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, που κερδίζουν τελικά πάρα πολλά χρήματα προωθούν ακριβώ αυτό το σύστημα καταβολής υποβολής προσφυγών. Προτεραιότητά μα θα πρέπει ανταυτού να είναι να διασφαλίσουμε την ευμερία και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών που μα εξέλεξαν, ενώ εσεί πρημοδοτείτε πάντα του λαθρομετανάστε κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Πέρα από την ανευθυνότητα αυτή είστε πραγματικά και ανήθικοι γιατί μας καλέσατε να πιούμε και σαμπάνια προκειμένου να γιορτάσουμε την έγκριση του νέου αυτού νομοθετικού κειμένου. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να λογοδοτήσει τα πέντε στους ίδιους τους πολίτες που σας εκλέγουν. Η κυρία Κίνιτσι για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό παρακαλώ. Κοιτάξτε, καλοδεχούμενοι οι επισκέπτες, αλλά εδώ μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, εκτός από το να χειροκροτάτε, εκτός από το να δείχνετε ότι συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καλό τους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου να παρέμβουν. Η κυρία Κινέση, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αυτό αφορά ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό χαρακτηρίζεται από πράξεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή και να υπάρξει βελτίωση της φιλοξενίας τους ε, σε όλους όσοι ζητούν άσυλο. Στο πλαίσιο λοιπόν των διατάξεων που ισχύουν είναι απαραίτητο να γίνονται έλεγχοι και οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνονται παράλληλα με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι το αντίθετο βοηθάει του διακινητές, όπω επίση και τη διάδοση άλλων μορφών οργανωμένου κλίματο συμπεριλαμβανομένου και τη συμπεριλαμβανομένη και τη τρομοκρατίας. Οι έλεγχοι πρέπει να συμβιβάζονται με πλήρη σεβασμό τη αξιοπρέπεια και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, για να μην ζήσουμε καταστάσει ε, όπω. Ε, η μετανάστες ε, να συνοστίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι προβλέπεται στο νόμο χωρίς να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια και όλα αυτά είναι παράτυπα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με βάση το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τις ελευθερίες των μεταναστών η μόνη που ξέρεις μπορεί να γίνει είναι σε ειδικέ περιπτώσεις. Εξάλλου θα πρέπει να αποφύγουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ε, μεταναστών που βρίσκονται σε καταβλισμούς ε, φιλοξενίας, ε, σε συνθήκες οι οποίες είναι παντελώς απαράδεκτες, κάτι που έχει επισημάνει και ο Ευρωπαίος Διαμασαλοβητής. Κατά την άποψή μου, μια ευρωπαϊκή εκτοφυλακή που θα συσταθεί θα πρέπει να ε, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους, έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή να εντοπίζονται οι τροτές ομάδες, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να καταστούν θύματα του οργανωμένου εγκλήματος. Ο κύριος Χένκελ, για να Κοιτάξτε, ως ε, μέλος της Amnesty International για πάρα πολλά χρόνια χάρηκα πάρα πολύ που έγινε σήμερα λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και είναι όνειδος ε, το πώς επιτίθενται πολλοί στη δική μου την πατρίδα κατά των προσφύγων και ε, βάζουν φωτιά και στα σπίτια τους. Προς όφελος όσων έχουν δικαίωμα να παραμείνουν σε μια χώρα πρέπει να μιλήσουμε και για τις υποχρώσεις τους. Οι πρόσφυγες οι οποίοι καταστρέφουν τα έγγραφά τους, τη ταυτότητάς τους ή αναφέρονται μεταφέρουν λάθος στοιχεία για την ταυτότητά τους. Εκείνοι οι οποίοι ε, θέλουν να μεταφέρουν τις διενέξεις, τις θρησκευτικέ και άλλες στην Ευρώπη θα πρέπει να αποστέλλονται πάρα αυτά στις πατρίδες τους. Και όσοι παραμένουν, για αυτούς πρέπει να ισχύει η ενσωμάτωση. Δεν είναι μόνο υποχρέωση των Ευρωπαίων, αλλά είναι υποχρέωση και των προσφύγων. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει κάποτε να εκπαιμφθεί από αυτό το κοινοβούλιο. Κύριε Χένκελ, κύριε Χένκελ, υπάρχει ε, μια ερώτηση από τον, τον κύριο Μπονάνο. Παρακαλώ κύριε Μπονάνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, εσείς είσαστε περισσότερο δημοκράτης από εκείνη που μίλησε προηγουμένως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε και θέλω να σας ρωτήσω, ε, θα συμφωνούσατε να υπάρχει ένα Γκουαντάναμο στην Ευρώπη. κύριος Χένκελ, κοιτάξτε, εγώ ε, μίλησα και ήμουν, όπως σας είπα, μέλος της ε, Διεθνούς Ήμουν σαφώς υπέρ της κατάργησης του Αγκαντάνομου. Τι να σας πω, προφανώς και όχι. Ο κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Στις εβδομάδες πληθαίνουν ανησυχητικά οι αναφορές διεθνών οργανισμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κακομεταχείριση μεταναστών και προσφύγων από τις αστυνομικές αρχές ανατολικοευρωπαϊκών κρατών μελών της ένωσης όπως και από τις αρχές της τουρκίας. η ευρωπαϊκή ένωση όμως οφείλει να υπερασπίζεται τις καταστατικές της αξίες δηλαδή τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και να καταδικάζει τις παραβιάσεις τους από οπουδήποτε και αν προέρχονται. δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες δεν είναι εγκληματίες αλλά εγκατέλειψαν την πατρίδα τους λόγω φόβου δίωξης ή αναζητώντας μια καλύτερη τύχη πρέπει να βρούμε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. και ακόμα η ένωση οφείλει να ρίξει όλο το βάρος της για να υπάρξει ειρήνη και ομαλότητα στην περιφέρειά της και ιδίως στη μέση ανατολή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο ώστε να σταματήσει η αναγκαστική προσφυγοποίηση των ανθρώπων. Ευχαριστούμε κύριε Κρυσόγονο. Η κυρία Άννα Γκόμες για δύο λεπτά. Ο πρόεδρο Τούσκ ντρόπιασε την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες ε, πηγαίνοντας ε, με κάτι που έμοιαζε με τον Ορμπάν μιλώντας ε, για το ότι δεν θα μπορούσαμε, λέει, να τους απορροφήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες αν συνεχίσουμε να αρνόμεθα, μιλώντας για ξένους μαχητές, ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις τρομοκρατικές επιθέσεις τελευταίες είναι Ευρωπαίοι και ότι οι πολιτικές μας μόνο έχουν επιδεινώσει τα Μόλεμπεκ, τα διάφορα Μόλεμπεκ και επίσης ε, ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών μας δεν μοιράζονται τις πληροφορίες και θέλουμε κράτη-μέλη όπως ε, το δικό μου που περιμένουν να δεχτούν τους πρόσφυγες ε, ενώ υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν καν να τους ε, δουν ε, και δυσκολεύουν τις διαδικασίες ασύλου. Δεν θα πάψουμε να δεχόμαστε έτσι μαζικά και ανεξέλεγκτα τους πρόσφυγες παρά μόνο εάν κάνουμε κάτι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία εκεί όπου πηγάζει. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές είναι να διοργανώσουμε με νόμιμες διόδους εισόδου της Ένωσης. Είναι πολύ πιο εύκολο να κόψουμε τα κέρδη των διακινητών. Όμως αυτά τις διόδους δεν τις υποστηρίζουν οι κυβερνήσεις μας. Δεν γίνεται να ελέγξουμε κάθε μέτρο ευρωπαϊκών συνόρων. Με όποιο... Το κόστος θα είναι τεράστιο. Απλώς θα τελειώσει έτσι το ευρωπαϊκό όραμα και θα παίξουμε το παιχνίδι των διακινητών και των τρομοκρατών. Δεν πρόκειται να σταματήσουν οι ροές, ούτε θα ε, νιώσουν δώσουν περισσότερη ασφάλεια οι πολίτες μας. Χρειάζεται ε, να ε, μοιραστούν τις πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και για να ε, μοιραστούμε την προσπάθεια υποδοχής για όσους μας δουν άσυλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασνοντιεύσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι μερικοί συνάδελφοι όταν μιλάνε για το νόμο και το δικαίωμα κατ' ουσίαν μιλάνε για αναρχία. Ε, χάνουν την αίσθηση της ε, πραγματικότητας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ερωτήσω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό τον μηχανισμό της μεταγκατάστασης, πώς τον φαντάζονται χωρίς να εφαρμόζεται βία. Μα πώς θα προβαίνετε στη δακτυλοσκόπηση η μετεγκατάσταση των προσφύγων δεν μπορεί να γίνει χωρίς δακτυλοσκόπηση. Οι ε, πρόσφυγες έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες όπου δεν επιθυμούν να ζήσουν. Όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, δεν θέλουν να ζήσουν ούτε στην Πολωνία, ούτε στη Λουθανία, αλλά στη Σουηδία και στην Πολωνία. Παρακαλώ, κυρία Τζούμπερ, για ένα λεπτό. Η χρήση βία κατά των ετούντων άσυλων είναι ντροπή, όπω είναι και η χρήση τη βία κατά των μεταναστών εν γέννη. Αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να χρησιμεύσει για να επιλέγουμε του ε, μετανάστες στην Πολωνία και στην ε, Βουλγαρία αλλά και στην Ουγγαρία. Είναι εντοπιστική κατάσταση. Όσοι διέσχισαν την Βουλγαρία χρειάστηκε να περάσουν διαπυρώσεις και σιδήρου μέσα από απάνθρωπε συνθήκε. Όμως επίσης η Τουρκία για παράδειγμα σπρώχνει με βία τους Σύριους πίσω στη Σύρια η Τουρκία, την οποία θέλει να δώσει δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει, υποτίθεται, τους, μετα, τους πρόσφυγες τους οποίους εκείνη απορρίπτει. Και στην Μεσόγειο ε, διώχθηκαν ε, πρόσφυγες. Ποιε είναι αυτέ οι δυνάμεις των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο κυριο Πόστα, για δύο λεπτά. Α, η κυρία με συγχωρείτε, κυρία Πόστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου κάνοντας μία αποτίμηση. Καταρχάς, κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί παράνομος μετανάστης. Η όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου θετική για τα άτομα στα οποία αναφερόμαστε. Τα όσα λέμε αυτή τη στιγμή για ανώτατα ωρία, για ποσότητες ανθρώπων οι οποίοι έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά δεν συνάδουν με την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θετικό παράδειγμα και θα πρέπει να λειτουργούμε απόλυτα λογικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίσουμε πώς μεταχειριζόμαστε τους μετανάστες αυτούς και όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μπορεί με στους μετανάστες να έχουμε ακόμα και εγκληματίες. Και βέβαια έχουμε και παράνομες περιπτώσεις διέλευσης των συνόρων, αλλά είναι ευθύνη των κρατών μελών να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στο εδαφός τους. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε βία ή να καταπατούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όταν αυτό γίνεται χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία είναι παράνομο να μην αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με αξιοπρέπεια ως ανθρώπινα όντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει λοιπόν μια πολύ σημαντική ευθύνη, έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν αυτή την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή επιτήρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε καλύτερα και τις προσφυγές που θα γίνονται πλέον από τους μετανάστες, ιδίως όταν καταπατώνται ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως πραγματικούς ανθρώπους. Διαφορετικά νομίζω ότι θα χάσουμε και εμείς την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. Ο κύριος Χουντής για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τούτο το χρόνο, το 2015, γιορτάζουμε τα 65 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό τη σκιά πολέμων, τρομοκρατίας και χιλιάδων προσφύγων η καταστολή η αστυνομική βία κατά των προσφύγων οι φράχτε, οι δημιουργία στρατόπεδα συγκέντρωση είναι ντροπή για την ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη τη παραπέμπουν σε άλλε σκοτεινέ περιόδου τη Ευρώπη που κανένα δημοκρατικό πολίτη δεν θέλει να αναβιώσει. το σύστημα του δουβλίνου παραβιάζει δικαιώματα χώρε όπω η ιταλία και η ελλάδα έχουν μετατραπεί σε αποθήκε ανθρώπων και το ερώτημα για το παρόν και το μέλλον της ευρώπης με τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν γίνεται όλο και πιο οδυνηρό. παραδείγματο χάρη η δημιουργία της νέας frontex εξασφαλίζει τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο. δεύτερο έναντι ποιου θα μπορούν να προσφύγουν όσοι αδικήθηκαν ή τους κακομεταχείρισαν. τρίτο πώς εξασφαλίζονται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. δυστυχώς η αλήθεια είναι τραγική η ευρωπαϊκή ένωση κινείται στα όρια του διεθνούς δικαίου μεταθέτοντας τις ευθύνες και στοχοποιώντα τα κράτη μέλη τη. οι πολιτικέ ευθύνε και οι ενοχέ τη ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορούν να καλυφθούν κατά την πίεση μικροπολιτικών συμφερόντων εθνικιστικών περιχαρακώσεων και ακραία ρητορική. ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε. Ξεκινάει τώρα η διαδικασία Catch the Eye. Πέντε ευρωβουλευτέ έχουν ζητήσει το λόγο. Γιάκοβιτ πρώτο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι μας έκανε σε όλους εντύπωση καταρχάς η προσφυγική αυτή κρίση και πολύ συχνά στα πλαίσια της κρίσης αυτής χρειάστηκε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα, αυθαίρετα και με έναν τρόπο μη συνεκτικό. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε ότι το σύστημα του Δουβλίνου δεν υφίσταται πλέον, δεν λειτουργεί στην πράξη. Είναι ανύπαρκτο το σύστημα αυτό. Έχει καταστεί αυτό σαφές. Σας το λέω αυτό, δεν ήμασταν έτοιμοι, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και τώρα από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την κατάσταση, ιδίω όσον αφορά τα σύνορα στην Ουγγαρία ή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα όσα συμβαίνουν στα σλοβενικά σύνορα, στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τις δηλώσεις του κυρίου Τούσκ, θεωρούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτες. Χώρες όπως η δεν μπορουμε να διαχειριστουμε τα οσα συμβαινουν στα σλοβενικα συνορα στα συνορα μεταξυ σλοβενιας και κροατιας δεν μπορουμε να αποδεχθουμε τις δηλωσεις του κυριου τους και θεωρουμε οτι ειναι εντελως απαραδεκτες χωρες οπως η Σερβία η πρώην Κωνσταντική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα πρέπει τρόπον την άνε υποστηριχθούν, γιατί θεωρώ ότι έχουν συμβάλει. Έχει κατακλειστεί από χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Πάνω από 500.000 πρόσφυγες έχουν εισέλθει στη χώρα μου. Το καλοκαίρι επισκέφθηκα τη Σάμο, την περασμένη Κυριακή την Ιδωμένη, στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Το Σάββατο θα επισκεφθώ τη Μυτιλίνη. Επομένως έχω εικόνα επιτόπια, on the spot, του τι συμβαίνει και σας λέω ότι ο φτωχοποιημένος από τα μνημόνια ελληνικός λαός έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για φιλοξενία των χιλιάδων προσφύγων. η κριτική που ακούστηκε για την ελλάδα είναι όχι μόνο άδικη αλλά και υποβολημιαία. συνάδελφοι ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών αυξήθηκε πολλαπλάσια από τη στιγμή που η κυρία μέρκελ κάλεσε τους πρόσφυγες στη γερμανία από τις 160.000 πρόσφυγες για μετεγκατάσταση έχουν προχωρήσει στη διαδικασία τα κράτη μόνο για 2.000 από τους μετανάστες και από τα 28 κράτη έχουν ανταποκριθεί μόνο τα 8. Επομένως, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους τα κράτη-μέλη της Ένωσης και ιδίως αυτά που ευθύνονται για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Eh, Υπάρχει λοιπόν ε, αυτή η συνεδρίαση ε, στην Ουγγαρία που, όπου έγινε λόγος για την προστασία των συνόρων. Για φανταστείτε ότι έχουμε μία επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση ε, είναι εγκατεστημένη σε ένα πολυτελές παλάτι και προσκαλεί μια αντιπροσωπεία. Έρχεται η αντιπροσωπεία και το Σαββατοκύριακο παρόν είναι μόνος, μόνο ο θηρορός. Και όταν όμως ε, μιλάει ο θηρορός με τους ιδιοκτήτες και τους λέει τι κατάσταση είναι αυτή, του λένε οι ιδιοκτήτες μη σας νοιάζει και μην στενοχωριέστε, πάρτε τους ε, στο σπίτι σπίτι σας, λένε στο θεωρό και φιλοξενήστε τους. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε με τους πρόσφυγες. Εσείς ε, με, με το αφεντικό σας, την κυρία Μέρκελ, εσείς οι Γερμανοί καλέσατε εκατομμύρια προσφύγων και τώρα θέλετε οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να φορτωθούν το πρόβλημα. Εμείς δεν το θέλουμε. Ο κύριος Τόμασίτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συστάμε το ζήτημα της μετανάστευσης ε, και των προσφύγων. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα και για τις υποχρεώσεις που έχουν οι μετανάστες, όχι μόνο τα δικαιώματα. Οι υποχρεώσεις είναι να τηρούν το Σύνταγμα και την νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται. Συντοπιώ πώς έχει η κατάσταση, συνειδητοποιώ ότι διαφεύγουν οι δεχθείς καταστάσεις, συμφωνώ ότι ορισμένοι να μην έχουν ακόμα ενσωματωθεί στην κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα, μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώ τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του. Νομίζω πάντω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε του μετανάστε με τρόπο ισότιμο, όπω αντιμετωπίζουμε και του πολίτε μα. Η δικαιοσύνη, ο νόμο θα πρέπει να είναι ο ίδιο για όλου. Ξέρω ότι η κατάσταση είναι κάπως χαοτική για τους ετούντες άσυλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναστείλουμε εμεί οι εθνικές μας νομοθεσίες ή ότι θα πρέπει να ανεχτούμε την μη τήρηση της δικής μας εθνικής νομοθεσίας. Όσοι θέλουν να ζήσουν στην Ευρώπη θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν να ενσωματωθούν στις δικές μας τις χώρες. Και η διαδικασία αυτή ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που θα πατήσουν πόδι στις χώρες μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα όσα ακούσαμε για την κράτηση των ετούντων άσυλο και για την χρήση βία για να καταγραφούν είναι ανησυχητικό. Εγώ επισκέφθηκα ένα κέντρο ε, αναγνώριση και ε, επαναπατρισμού στην Ιταλία. Δυστυχώ δεν τηρούνται τα δικαιώματά του μέσα, ούτε καν αυτό του να ζητήσουν άσυλο. Χωρίζονται και υπόκειται σε διακρίσει ανάλογα με την, την εθνικότητά του ανάμεσα στου κανονικού και αυτού που μπορούν να επιστραφούν. Μπορεί να κρατήσουν οι διαδικασίε μέχρι και ένα χρόνο. Οι συνθήκε διαβίωση στα κέντρα αυτά είναι χείριστε, υπάρχουν και ανήλικοι που δεν θα έπρεπε καν να είναι εκεί και η μέθοδο υπολογισμού του ε, ηλικία του με τον τον, ε, με την εξέταση του παλμού τους είναι ακατάλληλη τελείως. Ε, ε, θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε να τους δώσουμε τελικά μια σαφή προοπτική για το μέλλον τους. Γι' αυτό και το ξεπέρασμα του Δοφλίνου και το σχέδιο κατάσταση είναι πολύ καθυστερημένο και θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σλάιν και τώρα ολοκληρώνεται εδώ το Καρστιάι και τώρα τον λόγο θα πάρει ο Επίτροπος Στυλιανίδης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ καρποφόρα συζήτηση. Πολύ επικοδομητική και παραγωγική ήταν η συζήτηση. Γνωρίζετε ότι ο αγαπητός συνάδελφος Δημήτρης Αβραμόπουλος που είναι ο αρμόδιος για αυτό το θέμα στις συναρκτήριές του παρατηρήσεις ήδη κάλυψε όλες τις πτυχές αυτού του τόσο δύσκολου θέματος. Εγώ λίγα λόγια θα πω μόνο, ότι δηλαδή η Κομισιόν αναλαμβάνει δράση ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα του ασύλου. Το δικαίωμα του ασύλου είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και βεβαίως αυτό σημαίνει το σεβασμό όλων των πτυχών της νομοθεσίας περί ασύλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν στη διάρκεια του περασμένου εξαμήνου έχει στείλει τρεις αιτιολογημένες θέσεις 42 επιστολές επίσημες κοινοποίησης και 8 διοικητικές επιστολές στον τομέα της, του ασύλου όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού Eurodac και επίσης τη μεταγραφή της συμμόρφωσης όσον αφορά τις οδηγίες για το άσυλο. Θα ήθελα να τονίσω και να εστιάσω σε αυτό ότι το δικαίωμα στο άσυλο είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα και βεβαίως αυτό σημαίνει σεβασμό όλων των πτυχών της νομοθεσίας περί ασύλου. Στην, η Κομισιόν παραμένει απόλυτα προσιλωμένη στην εξασφάλιση του σεβασμού από πλευρά των κρατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όταν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε και τώρα δίνω αμέσω το λόγο στον Υπουργό Σμίτ εξ του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, Ευρωβουλευτές, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εγώ να πω ότι ε, μπορώ να ερμηνεύσω ότι εκπροσωπώ αναγκαστικά τα όσα έχει πει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάντως διαβάζω εδώ πέρα την επιστολή την οποία έστειλε προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Αυριανό και σας διαβάζω τι λέει στα αγγλικά η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων δεν έχει ως στόχο να φοβήσει αυτούς οι οποίοι διαφεύγουν πολέμους ή διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει πάντα υποδοχή σε όλους αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν. Όπως και Επίτροπος, έτσι και εγώ είπα, ποια είναι η νομοθεσία όσον αφορά την κράτηση των ετούντων άσυλο. Η κράτηση λοιπόν των ετούντων άσυλο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή να προσεγγιστεί αποκλειστικά ως κανόνας ή ως ομοναδικός κανόνας αν υπάρχουν καταχρήσεις, αν υπάρχουν καταστάσεις όπου οι ευρωπαϊκοί κανόνες ή οι διεθνοί κανόνες δεν τηρούνται, τότε θα πρέπει να αναλάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, γιατί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ατιμωρητοί να παραβιάζονται. Ακριβώς λοιπόν επειδή αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση κρίσης αυτή τη στιγμή, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο θεωρώ να ξαναδιαβάσουμε τα θεμελιώδη κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα οποία καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι, ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Τα κείμενα λοιπόν αυτά, μεταξύ άλλων είναι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο πρώτο άρθρο του χάρτη αυτού, στο πρώτο άρθρο του χάρτη αυτού λέγεται το ακόλουθο λέγεται ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να παραβιάζεται, ότι θα πρέπει να τηρείται και να προστατεύεται σε κάθε περίπτωση. Και στο άρθρο 18 της χάρτας λέγεται ότι το δικαίωμα ασύλου προασπίζεται από τη Σύμβαση της Γενέβης και από άλλα διεθνή κείμενα. Αυτές είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές μας και προφανώς όλοι θα πρέπει να τηρούν τις εθνικές νομοθεσίες, τους εθνικούς κανόνες και βέβαια εκεί αιτούνται σε άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση.